Dobrý den, dámy a pánové. Já vás vítám na našem dnešním Καλημέρα σα αγαπητοί συνάδελφοι. Καλώ ήρθατε στη σημερινή συνεδρίαση. Ήθελα να καλωσορίσω του ε, προσκεκλημένου μα, Περνάει η ώρα, γι' αυτό ας εγκρίνουμε την ημερήσια διάταξη. Δεν νομίζω πω υπάρχει κάποια αντίρρηση επί τη ημερήσια διάταξη. Εγκρίνεται λοιπόν. Επίσης, εγκρίνονται και τα πρακτικά, αφού δεν υπάρχει κάποια αντίρρηση. Θα αρχίσουμε λοιπόν ευθύς αμέσως. Θα ήθελα να καλωσορίσω τον προσκεκλημένο μας κύριο μάθια Υποπόφσκι, αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης. Θα μας μιλήσει για ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Και αμέσως μετά την παρουσίαση του κυρίου Ποπόφσκι θα γίνει ανταλλαγή απόψεων. Και μια που έχουμε αργήσει πάρα πολύ, θα ήθελα να σας παρακαλέσω να είστε πειθαρχημένοι στο χρόνο ομιλία σας. Κύριε Παπόφσκι, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Συνεδρίασαν αρχικά οι Υπουργοί Άμυνας και μετά οι Υπουργοί Εξωτερικών στις 18 Μαΐου λοιπόν. Κύριο θέμα του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων ήταν η προετοιμασία των συζητήσεων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για την Ασφάλεια και την Άμυνα. Συζητήθηκαν όμω και άλλα πράγματα πέρα από αυτά, διότι η επιθυμία ήταν να δημιουργηθεί μια θαλάσσια επιχείρηση στη Μεσόγειο, η οποία και δημιουργήθηκε εκείνη την ημέρα. Θα επανέλθω όμως από αυτού. Είπατε εκπρόσωπος, κυρία Μοκερίνη, συμμετείχε στις συζητήσεις για το άρθρο 36 και αναφέρθηκε σε πολλά θέματα της ημερήσιας διάταξης στο Υπουργικό Συμβούλιο. Η συνεδρίαση άρχισε με την Δικούσα Επιτροπή για την Άμυνα. Συζητήθηκε η πρόοδος στην ανάπτυξη δυνατοτήτων. Και έπειτα συζητήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και η προετοιμασία για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Είπα ότι εκπρόσωπο συμμερίστηκε την άποψη των Υπουργών Άμυνα ότι δηλαδή υπάρχει επιθυμία να δημιουργηθεί σωστή ε, ε, ισορροπία ανάμεσα στην εφαρμογή των αποφάσεων του 2015 και των στόχων για το μέλλον, των προτεραιοτήτων δηλαδή για τα επόμενα χρόνια. Το σκεπτικό ήταν πώς η ασφάλεια και η άμυνα να παραμείνει στην ημερήσια διάταξη των ε, αρχηγών κυβερνήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό λοιπόν πιστεύω πως το Συμβούλιο του Ιουνίου δεν θα είναι απλά διεκπαιρεωτικό, αλλά θα συζητηθούν ορισμένοι τομεί προτεραιότητα, στους οποίους θα δοθεί έμφαση μετά τον Ιούνιο του 2015. Τώρα δεν θα σας απασχολήσω πολύ με τις επιχειρήσεις. Υπήρξε μια ενημέρωση για την ε, ισχύουσα κατάσταση των στρατιωτικών επιχειρήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρουσιάστηκαν πέντε από αυτές από τον πρόεδρο της Στρατιωτικής Επιτροπής. Και έπειτα η, ε, στους υπουργούς προσθέθηκε και ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ για να συζητηθεί το περιβάλλον ασφαλείας στη Νότια και Ανατολική Μεσόγειο ήταν ευπρόσδεκτος ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, διότι φυσικά όλοι έχουν κοινούς στόχους και κοινή τακτική για πολλά από τα θέματα. Και είπατε εκπρόσωπος λοιπόν και ο Γενικός Γραμματέας δεσμεύτηκαν να βελτιωθεί όσο το δυνατόν περισσότερο η σχέση Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΝΑΤΟ. Τώρα, όσον αφορά τι προετοιμασίε για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, ε, καλύφθηκε η δημιουργία δυνατοτήτων. Το δεύτερο σημείο δηλαδή τη δική σα σημερινή ημερήσια διάταξη. Δεν θα μπω λοιπόν σε λεπτομέρειε από τώρα. Ε, ήταν μια πρωτοβουλία η οποία ονομαζόταν Train and Equip, κατάρτιση και εξοπλισμός. Τώρα έχει μετονομαστεί για την, ε, σε δημιουργία δυνατοτήτων σε τρίτες χώρε. Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε πριν από μερικές εβδομάδες ένα σχετικό έγγραφο πολιτικής το οποίο θα συζητήσουμε αργότερα μαζί με τον συνάδελφό μου Μάρκος Κορνάρα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι υπουργοί συζήτησαν ζητήματα των ε, αμυντικών δαπανών. Θεωρείται πως πρέπει να σταματήσει η περαιτέρω μείωση των αμυντικών δαπανών. Οι συγκεκριμένοι αμυντικοί στόχοι αναφέρθηκαν και από το ΝΑΤΟ και επιβεβαιώθηκαν στην διάσκεψη στη Σύνοδο της Ουαλίας. Αποφασίστηκε λοιπόν ότι για να βελτιωθεί ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα κονδύλια χρειάζονται νέες μέθοδοι αντιμετώπισης, νέες προτάσεις. Υπήρξαν κάποιες προτάσεις που υποβλήθηκαν και σχετικά με την εξοικονόμηση πόρων και με τη βελτίωση των, ε, του τρόπου που δαπανώνται οι φυσταμένοι πόροι. Η συνεισφορά είναι ακόμα εθελοντική. Η πολιτική, η αμυντική πολιτική είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών, όμως υπήρξε επιθυμία τα κράτη να συνεργάζονται μεταξύ τους και σε αυτό επετέφθη πρόοδος. Υπήρχαν κάποιες εξαιρέσεις στο θέμα του ΦΠΑ που χορηγήθηκαν σε ορισμένα προγράμματα για το Βέλγιο για παράδειγμα και διερευνάται το ενδεχόμενο ενός υποστηρικτικού μηχανισμού ή κάποιου αμυντικού ταμείου το οποίο θα αναλάβει συντονιστικό ρόλο στον προϋπολογισμό για την άμυνα. Προσπαθούμε λοιπόν να συγχρονιστούμε και να συντονίσουμε καλύτερα τις αμυντικές δαπάνες. Συζητήθηκαν έπειτα οι προπαρασκευαστικές δράσεις για την ε, κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας. Το νέο πρόγραμμα θα τεθεί σε ισχύ επίσημα το 2017 και ο προϋπολογισμός θα είναι ο πρώτος ευρωπαϊκός προϋπολογισμός για την έρευνα και την ανάπτυξη στην πολιτική ασφάλειας και άμυνας. Τα κονδύλια αυτά δεν θα δαπανηθούν στην απόκτηση αμυντικών συστημάτων, αλλά όπως και στα πλαίσια του ορίζοντας 2020, ε, σε έρευνα και ανάπτυξη που σχετίζεται με στρατιωτικά και αμυντικά ζητήματα. Έχει οριστεί μια ομάδα εμπειρογνωμόνων η οποία θα έχει συμβουλευτικό ρόλο και θα συμμετέχει στην προπαρασκευαστική φάση του προγράμματος εν του νέου πολίτου δημοσιονομικού πλαισίου. Η ομάδα αυτή η εμπειρογνωμόνων θα αποτελείται και από πολιτικούς και από εκπροσώπους της ε, βιομηχανίας και από, το, από εκπροσώπους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Έχουν ήδη αναλάβει τις αρμοδιότητές τους, έχουν ήδη αρχίσει να εργάζονται και την άνοιξη του 2016 θα δημοσιευτεί η τελική τους έκθεση. Επίσης, οι Υπουργοί τόνισαν τη σημασία της ε, πιο εύκολη ε, πρόσβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην αγορά αμυντικών συστημάτων. Συζητήθηκαν επίσης οι νέες μορφές απειλής, υβριδικές απειλές. Υπήρξε δέσμευση να υποβληθούν νέες προτάσεις κατά τη διάρκεια του έτους για το πώς θα αντιμετωπιστούν αυτές οι υβριδικές απειλές, σε συνεργασία βέβαια με το ΝΑΤΟ, το οποίο θα δώσει μια διαφορετική διάσταση στο θέμα, διότι για το ΝΑΤΟ οι υβριδικές απειλές ε, σημαίνουν κυρίως σχεδιασμό και πρόβλεψη και την αντιμετώπιση των ε, νέων συνθήκων που έχει επιφέρει η πρόοδος της τεχνολογίας. Επίσης, η ΥΠΑΤΗ εκπρόσωπος ενημέρωσε σχετικά με την στρατηγική αναθεώρηση μετά από το Συμβούλιο του 2013, η οποία θα οδηγήσει στην έγκριση της νέας στρατηγικής. Πρώτο στάδιο είναι η αξιολόγηση της στρατηγικής έκθεσης η οποία θα παρουσιαστεί στο Συμβούλιο του Ιουνίου. Είναι σχεδόν έτοιμη. Και η πλήρη στρατηγική θα παρουσιαστεί το 2016. Είπατε εκπρόσωπος αναφέρθηκε στην άνοιξη του 2016 ως μια ημερομηνία. Θέλει να γίνει ανταλλαγή απόψεων με όλους τους ενδιαφερομένους φορείς, και με την πανεπιστημιακή κοινότητα επίσης. Η μέθοδος είναι η ίδια με εκείνη που χρησιμοποίησε και ο Χαβιέ Σολάνα στο παρελθόν όταν δημιουργήθηκε πρώτη φορά η κοινή ευρωπαϊκή στρατηγική. Επίσης τίθηκε και η ε, απάντηση στην μεταναστευτική κρίση που έχει προκύψει. Όπως ξέρετε, η ατζέντα που έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη μετανάστευση έχει εγκριθεί περιλαμβάνοντας και πολλές ακόλουθες δράσεις σχετικά με την ε, επανεγκατάσταση προσφύγων. προβλέπονται επίσης και δράσεις στη θάλασσα που θα στοχεύουν στην ε, καταπολέμηση των διακινητών στη Μεσόγειο. Η απόφαση για να δημιουργηθεί αυτή η ομάδα ελήφθη το Μάιο, κάτι που ήταν αρκετά γρήγορο για τα ευρωπαϊκά δεδομένα. Η επιχείρηση λοιπόν αυτή δημιουργήθηκε ορίστηκε η έδρα στη Ρώμη της επιχείρησης αυτής και επικεφαλής ετέθη ένας Ιταλός ναύαρχος. Και αν πάνε όλα καλά, η επιχείρηση αυτή θα τεθεί σε ισχύ πολύ σύντομα, τους επόμενους μήνες. Φυσικά αναμένουμε και τις συζητήσεις στη Νέα Υόρκη και τα αποτελέσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας πρωτού αρχίσει η ανάπτυξη των δυνάμεων. Όμως είδαμε μεγάλη θέληση και νομίζω πως όλα θα πάνε όπως προβλέψαμε. Επίσης αναμένεται και η συμφωνία της ε, κυβέρνησης της ε, Λιβύης για την ανάπτυξη αυτή των ε, θαλάσσιων επιχειρήσεων στη Μεσόγειο. Φυσικά ξέρετε πως υπάρχουν δύο κυβερνήσεις στη Λιβύη αυτή τη στιγμή και είναι κάπως δύσκολη η συνεννόηση. Μία κυβέρνηση στην Τρίπολη, μία άλλη στο Τομπρούκ. Υπάρχουν λοιπόν δυσκολίες στο συντονισμό για την καταπολέμηση των διακινητών και κάποια προβλήματα όσον αφορά την ανάπτυξη επιχειρήσεων διάσωσης και εντοπισμού. Και μην ξεχνάμε ότι οι πρόσφυγες αυτοί πρέπει να απολαμβάνουν όλα τους τα δικαιώματα όπως προβλέπεται από Σύμφωνο της Γενέβης. Τέλος. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ιουνίου θα ασχοληθεί με δύο-τρία πολύ σημαντικά θέματα. Την ε, στρατηγική αναθεώρηση, όπως σας είπα, όπου αναμένεται να συζητηθούν τα χρονοδιαγράμματα και η ανάγκη ενός σταθερού πλαισίου. Οι επιχειρήσεις, όπως σας είπα, οι προπαρασκευαστικές δράσεις που θα προωθήσουν την συνεργασία σε αμυντικά ζητήματα στην Ευρώπη. και έπειτα η ανάμειξη των ενδιαφερόμενων φορέων στην ε, κατάρτιση και την δημιουργία δυνατοτήτων. Κάτι που θα συζητήσουμε σε λίγο. Θα σταματήσω λοιπόν εδώ κύριε Πρόεδρε, αλλά με τα χαρά να απαντήσω σε όποιες ερωτήσεις έχετε. Σας ευχαριστώ κύριε Ποπόφσκι για την ε, πολύ συνολική σας ε, επεξήγηση. Πριν αρχίσει η συζήτηση θα ήθελα να σας ειδοποιήσω ότι η επόμενη συνεδρίασή μας στις Σέτε στις 17 Ιουνίου εκεί θα έχουμε την Επιτροπή Γιανκόφσκα. Πριν από την συζήτηση θα ήθελα να ρωτήσω εγώ ο ίδιος κάποια πράγματα. Αναφερθήκατε στον υβριδικό πόλεμο. Επανειλημμένα ε, και σε συναντήσεις με φίλους και στην Επιτροπή τα έχουμε συζητήσει αυτά. Ε, πρόκειται για υβριδικό πόλεμο με την έννοια ανάμεσα από τον ψυχρό και τον θερμό πόλεμο ε, πρόκειται για κυβερνοεπιθέσεις. Και, εν πάση περιπτώσει, θεωρείται ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σε υβριδικό πόλεμο ε, με ή εναντίον της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Αυτή είναι η πρώτη μου ερώτηση. Η δεύτερη ερώτηση. Η έκθεση της ρωσικης ε, ομοσπονδιας αυτη ειναι η πρωτη μου ερωτηση δευτερη ερωτηση η εκθεση της της υπάτου του ε, εκπροσώπου άλλαξε. Μάλλον ε, ε, αναφέρει ότι πιάστηκε εξαπίνες κατά κάποιο τρόπο η Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά την ασφάλεια και την άμυνα. Θεωρείτε ότι οι κύριες αλλαγές τα τελευταία δύο-τρία χρόνια αυτές οι αλλαγές τις οποίες ε, πρέπει να αντιμετωπίσουμε και να προετοιμαστούμε να τις ε, ε, αντιμετωπίσουμε είναι τόσο σοβαρές. Αυτές είναι οι ερωτήσεις μου και θα ήθελα τώρα να ξεκινήσει η συζήτηση. Πρώτος ο κύριος Ντονζόν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ζητώ συγγνώμη γιατί δεν ήμουν από την αρχή της παρέμβασής σας και επομένως δεν ξέρω εάν θίξατε το συνολικό ζήτημα της χρηματοδότησης, ιδιαίτερος δε δύο σημεία, τα οποία συζητήθηκαν στο Συμβούλιο του Δεκεμβρίου 2013 και είχαν, ε, είχε, είχαν γύρει κάποιες ε, ε, ελπίδες, κυρίως όσον αφορά τον μηχανισμό Αθήνα. Ε, συζητήθηκε το θέμα αυτό σε επίπεδο υπουργών ή όχι. Και επίσης θα εγγραφεί το, στο επόμενο Συμβούλιο των Ιουνίου. Και κάτι άλλο πολύ σημαντικό, ε, ε, τα κίνητρα, κυρίως δε τα φορολογικά κίνητρα. Ενδεχομένως βέβαια αυτό αφορά περισσότερο την Κομισιόν, αλλά έχετε να μας πείτε κάτι όσον αφορά τα φορολογικά κίνητρα τα οποία θα μπορούσαν να δοθούν κυρίως ε, όσον αφορά τις αγορές από κοινού ε, ικανοτήτων μέσα από ευρωπαϊκό διάβλο. Το δεύτερο σημείο. Ε, θα ήθελα να επανέλθουμε στην απάντηση που δίδεται ε, στο στρατηγικό σκέλος στο πρόγραμμα της μετανάστευσης. Μίλησα σχετικά στην Ολομέλεια την προηγούμενη εβδομάδα και εξέφρασα μεγάλο σκεπτικισμό όσον αφορά το θέμα αυτό. Πιστεύω ότι αυτή η ναυτική στρατιωτική επιχείρηση δεν μπορεί να δώσει την προσήκουσα απάντηση. Άλλωστε υπάρχουν και ε, νομικά προσκόμματα τα οποία αναφέρατε. Αποσιωπούμε τα επιχειρησιακά προσκόμματα γιατί ακόμα προσωπικά δεν ξέρω πώς μπορούμε ε, ε, να διαλύσουμε, να καταστρέψουμε πλοία. Ε, το πώς μπορούμε να καταστρέψουμε πλοία στο πέλαγος ε, αφού τα έχουμε αδειάσει από τους ε, μετανάστες, ναι, αλλά πριν ξεκινήσουν, πριν ξεκινήσουν το ταξίδι τους, όσο βρίσκονται ακόμα αραγμένα στη Λιβύη, δεν μπορώ να το καταλάβω. πραγματικά δηλαδή από τη στιγμή που σε πραγματικό χρόνο θα μας δοθεί η πληροφορία, μέχρι τη στιγμή που θα προχωρήσουμε επιχειρησιακά στην καταστροφή αυτού του πλοιαρίου, δεν κατανοώ πώς θα γίνει η διαδικασία. Επίσης, ε, στρατιωτικές ε, αεροπορικές επιδρομές και χτυπήματα ε, τα οποία μπορεί να έχουν πολλέ, πολλά Je pense on va Πολλά παράπλευρα θύματα και καταστροφές επίσης δεν καταλαβαίνω πώς θα μπορούσαν ε, να γίνουν. Πιστεύω ότι οι πολιτικές ε, αποφάσεις ελήφθησαν πάρα πολύ γρήγορα, πρωτοφανές για την ε, πολιτική ασφάλειας και άμυνας, αλλά επιχειρησιακά εξακολουθούν να υπάρχουν πολλά προβλήματα κατά την δική μου προσωπική άποψη. Ε, βλέπω μεγάλη εφορία και μεγάλη χαρά και απλότητα στην όλη συζήτηση, λες και όλα θα μπορούσαν να γίνουν πάρα πολύ απλά. Αναρωτιέμαι, δεν θα μπορούσαμε να ανοιχνεύσουμε άλλες μορφές παρέμβασης, λιγότερο θεαματικές ενδεχομένως, λιγότερο λιγότερο εύκολες να τις πουλήσει κανείς εντός εισαγωγικών στο κοινό. Ε, δεν θα μπορούσαμε λοιπόν να προβλέψουμε ας πούμε πολιτικές αποστολές για τις χώρες διαμετακόμισης, κυρίως την, ε, τον Ήγυρα. Βλέπουμε ένα τρίτο των, ε, των μεταναστευτικών ροών έρχεται από την Ασία, ένα τρίτο από το κέρας της Αφρικής, ένα τρίτο από την υποσαχάρια Αφρική περνώντας μέσα από, τις, ε, το Σαχέλ και ε, από τον Νίγηρα κλπ. Φτάνοντας στη Λιβύη, στον Νίγηρα, έχουμε ήδη επιτόπου μία αποστολή η οποία θέλει να βοηθήσει ε, την Εθνική Φρουρά, το στρατό, την αστυνομία και τα τελωνία. Δεν θα μπορούσαμε να διευρύνουμε λίγο, να ισχυροποιήσουμε κατά κάποιο τρόπο αυτή την αποστολή έτσι ώστε να κάνει ε, και επιχειρήσεις ε, κατά της, ε, των μεταναστευτικών ροών. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι και στο Μαλί και στην Μπουρκίνα Φάσο και στην, στον Νίγηρα υπάρχει μεγάλη διαφορά της ε, ε, όλου του κυβερνητικού μηχανισμού που βοηθάει τη διαμετακόμιση αυτή των μεταναστευτικών ροών. Το λέω γιατί όταν φτάνουν οι μετανάστες πλέον στη Λιβύη είναι πια αργά. Δεν θα μπορούσαμε στην αρχή της αλυσίδας, σε χώρες όπως ο Νίγηρας και το Μαλί, όπου έχουμε ήδη επιτόπου αποστολές. Ξέρω ότι στο Κόξ έγινε λόγος γι' αυτό. Ε, δεν θα μπορούσε να συζητηθεί και στο, σε επίπεδο πολιτικών ε, και υπουργών, έστω και αν δεν είναι τόσο ελκυστική και σεξι αυτή η προοπτική και σίγουρα λιγότερο θεαματική. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Ντοζό. Θα ήθελα θα ήθελα να αναφερθώ κι εγώ σε κάτι αντίστοιχο. Ενδεχομένως οι τρίτες χώρες με την ε, συμμετοχή των τρίτων χωρών. Δεν θα μπορούσαμε ενδεχομένως σε κάποιες χώρες να δημιουργήσουν κάποιους χώρους υποδοχής των μεταναστών στον Νίγηρα Φερρυπίν ή κάπου αλλού. Ο κύριος Μπόντεν. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Για την, αυτό τον υβριδικό πόλεμο που αναφέρατε. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε εδώ όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων και επιχειρήσεων τύπου κλασικής ΚΑΓΕΒΕ της ε, Σοβιετικής Ένωσης δολοφονίες σκάνδαλα ιστορίες του τύπου υποστήριξη πολιτικών κομμάτων διαδηλώσεις όλα αυτά και μετά φτάνουμε σε ένα πιο ε, έντονο φάσμα δραστηριοτήτων ε, και μοντέρνο. Κυβερνο επιθέσεις, τέτοιου είδους ε, δραστηριότητες. Θα πρέπει να συνειδητοποιούμε ότι ο, σε οποιοδήποτε από αυτούς τους τομείς μπορεί να υπάρξει πρόβλημα. Ξέρει ο κύριος ε, πόσο σημαντική βρίσκω ότι είναι η κοινωνική μας πολιτική, αλλά χαίρομαι που φίλος και συνάδελφος κύριος Ντονζό εκφράζει τον σκεπτικισμό του όσον αφορά το τι έχει να κάνει εδώ το θέμα Τώρα, ποιος είναι ο κύριος στόχος στα πλαίσια του Συμβουλίου τον Ιούνιο. Τι πιστεύετε ότι θα αποφασίσει. Ποιο θα είναι το διατάφτα. Τώρα σαν αφορά την ε, νέα αυτή πολιτική που θα δημιουργήσουμε στη Ρώμη από την, ε, στην κοινότητα για να αντιμετωπίσουμε αυτά τα προβλήματα. Επισκέφθηκα ε, εγώ τις κατάσταση, Πρόκειται για μία ε, στρατιωτική ε, βάση Ιταλική θα υπάρξει κοινοτική δράση, θα υπάρξει προσωπικό ώστε αυτή η η Ιταλική βάση να αποτελέσει την έδρα των επιχειρήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην ε, σχετική συνεδρίαση που έγινε θεωρήθηκε ότι θα μπορούσε να υπάρχει ε, μία ρύθμιση τύπου Βερολίνο Plus. Ξέρουμε ότι υπάρχει και στην Άπολη για θέματα ε, εποπτείας και στρατιωτικών επιχειρήσεων στην περιοχή της Μεσογείου και η έδρα του ΝΑΤΟ εκεί. Όπως επίσης σωστά ανέφερε ο κύριος Ντόζο, η στρατιωτική δράση. Στη νέα αυτή επιχείρηση έχουμε να κάνουμε με τον διακίνηση, παράνομη διακίνηση των μετανοστών. Δεν έχει καμία σχέση με τις κανονικές ροές μετανοστών. Και βεβαίως δεν πιστεύει κανείς ότι θα στείλουμε όλο μας το ναυτικό στόλο στην Ευρώπη για να σταματήσουμε τους πάντες. Το είπε ο κύριος Δονζό. Χρειαζόμαστε να δούμε πώς δημιουργήθηκε το όλο πρόβλημα και να αναλάβουμε δράση ευθύ εξ αρχής, ώστε να εμποδίσουμε τα άτομα αυτά να φτάνουν στις ακτές ε, της Αφρικής προς την Ευρώπη. Και βεβαίως η Ερυθρέα είναι μία από τις ε, περιοχές στις οποίες γίνονται διάφορα πράγματα δίπλα στο Τζιμπουτί. Διερωτώμε με, στο Τζιμπουτί ξέρει κανείς τι γίνεται στη γειτονική τους χώρα, την Ερυθρέα. Γιατί φτάνουν εκεί όλα αυτά τα άτομα και με ποιο τρόπο. Διερωτώμε λοιπόν, ποιες προσπάθειες θα γίνουν ώστε να μπορέσει και να ενισχυθεί ο επαναπατρισμός των μεταναστών. Διότι Αυτό το οποίο ε, πιστεύουν κάποιοι είναι ότι όταν φτάσει στην ε, ακτή έχουν δει τα προβλήματά του. Θα πρέπει αυτή η άποψη να αλλάξει. Δεν μπορούμε να τους στέλνουμε σε όλες τις χώρες και να νομίζουν ότι έχουν τα προβλήματά τους και βεβαίως και στη δική μου. Και εμείς όπως ξέρετε έχουμε έναν συντηρητικό πρωθυπουργό στη Μεγάλη Βρετανία που τέτοιου είδους μέτρα θα τα αρνηθεί. Πιστεύω λοιπόν ότι πρέπει να κάνουμε σε αυτή την κατεύθυνση κάτι και να λάβουμε μέτρα. Να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή και όχι να τα αφήσουμε όλα να γίνουν στα πλαίσια της κοινή πολιτικής στην Ευρώπη, έτσι όπως προβλέπετε στην ε, συνεργασία. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Σιμπάης. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ξεκινήσω λέγοντας ότι συμφωνώ απολύτως με όσα είπε ο κύριος Ντανζόν αναλύοντας ε, την ε, νέα στρατηγική επιχείρηση για την οποία ελήφθη απόφαση στο Συμβούλιο των Υπουργών. Είναι παράλογη αυτή η απόφαση. Δεν, δεν μπορεί να βασιστεί σε καμία πραγματικότητα. Ε, ε εμείς ήρθαμε σε επαφή και ακούσαμε τον Πρωθυπουργό της Τινησίας ο οποίος σαφέστατα αντιτίθεται σε αυτήν την πρόταση και θεωρεί ότι δεν μπορεί να λυθεί το πρόβλημα της μετανάστευσης με αυτόν τον τρόπο. Ε, αλλά λάβαμε και ε, μία επιστολή από τον ε, εκπρόσωπο πρέσβη της Λιβύης, της κυβέρνησης με την οποία εμείς έχουμε επαφές, που επίσης αντιτίθεται. Η κυρία Μογκερίνη προσπαθεί να πείσει όλο τον κόσμο ότι πρέπει να υπάρξει οπωσδήποτε μία, ένα ψήφισμα από πλευρά των εθνών έτσι ώστε να επιβεβαιωθεί η παρέμβαση. Ε, προσπαθούμε ε, να ε, έχουμε ένα ψήφισμα στο Συμβούλιο Ασφαλείας αλλά θα πρέπει, του, του αυτό θα πρέπει να γίνει απλώς για να μπορέσει να σταματήσει η κατάσταση στην Λιβύη και να μπορέσουμε να περάσουμε στο επόμενο βήμα. Με κανένα τρόπο αυτό δεν θα αποτελέσει λύση για το μεταναστευτικό πρόβλημα. Ε, όσον αφορά τώρα τις απειλές ε, προς την ασφάλεια, ε, κοιτάξτε, πολύ συχνά οι μετανάστες θεωρούνται ένα, μια τέτοια απειλή. Εγώ δεν νομίζω ότι απειλή είναι οι μετανάστες. Απειλή για την ασφάλεια βρίσκεται στις χώρες από τις οποίες ξεκινούν αυτοί οι μετανάστες. Οι ίδιοι οι μετανάστες, οι ίδιοι οι άνθρωποι δεν απειλούν την ασφάλεια. Τώρα, τα, ε, στα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 18ης Μαΐου αναφέρεται ότι ε, θέλουμε να ζητήσουμε επισταμένως ε, μία δράση από πλευράς ΕΕ και κρατών μελών. Αλλά εάν δεν κάνω λάθος... Οι χρηματοδοτήσεις των κρατών μελών προς τα Ηνωμένα Έθνη έχουν μειωθεί ε, και η δέσμευση επίσης στα πλαίσια των αποστολών των Ηνωμένων Εθνών, η δέσμευση ο πλευράς κρατών μελών επίσης ε, έχει μειωθεί. Ε, γίνεται λόγος ε, και για ένα γενικότερο ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Πάντως εγώ νομίζω ότι θα πρέπει να πούμε ότι ίσως, ίσως καλύτερα θα, έχουμε, θα, ήταν να έχουμε ένα ρυθμιστικό πλαίσιο ε, έτσι ώστε να ξέρουμε τουλάχιστον για τα drones, για τα μη επανδρομένα αεροσκάφη, να ξέρουμε ακριβώς τι θα κάνουν. Τώρα, ε, μιλάμε για την ε, ε, βιομηχανία των όπλων και την βλέπουμε σαν πάροχο θέσεων, θέσεων εργασίας. Όμως ξεχνάμε γιατί υπάρχει αυτή η βιομηχανία. Η, η, κύρια βιομηχανία, ο κύριος λόγος συγγνώμη, για τον οποίο έχουμε βιομηχανία εξοπλισμών στην Ευρώπη είναι έτσι ώστε να έχουμε μια βιομηχανία η οποία να μπορεί να βοηθεί λύση στην ασφάλεια της ε, χώρας μας. Θα πρέπει να δούμε τι γίνεται και με τις εξαγωγές όμως που κάνει ενδεχομένως αυτή η βιομηχανία μας γιατί μέσω των εξαγωγών έχουμε εν μέρη συμβάλει ε, στους πολέμους ε, σε διάφορα σημεία του κόσμου και στην κατάσταση η οποία έχει, υπάρχει πλέον στην Μέση Ανατολή και πιο πέρα. Θα πρέπει να τα δούμε όλα αυτά τα πράγματα με καθαρό βλέμμα. Ευχαριστώ πολύ κυρία Σαβάγιος. Κύριο αν έχει το λόγο, αλλά θα ήθελα να ερωτήσω το εξής. Όλοι ξέρουμε ότι εσείς είστε ε, εμπειρογνώμων σε θέματα που αφορούν τη Ρωσία. Μπορείτε να μας πείτε δεδομένου ότι σε θέματα ασφαλείας ε, επειδή είναι χώρα γειτονία προ την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι σημαντική η Ρωσία. Τι μπορεί να μας πείτε για τη Ρωσία σε αυτή την περίπτωση. Διαδικαστικό. Υπάρχει κάποιο πρόβλημα ίσως που δημιουργήθηκε από την ε, ε, διερμηνία ε, έχουμε την αμυντική βιομηχανία γιατί χρειαζόμαστε προστασία και όχι για να δημιουργούνται θέσει απασχόλησης. Μάλλον στη γραπτή μετάφραση λέει ο Μιλήτρη υπάρχει κάποιο λάθος, κάποια παρανόηση. Παρακαλώ να διορθωθεί. Σας ευχαριστούμε για την παρατήρησή σας, τη λαμβάνουμε υπόψη. Αγαπητέ Πρόεδρε, πολλές ικανότητες που ίσως δεν διαθέτω μου αποδίδεται. Εν πάση περιπτώσει. Την πρώτη ερώτησή μου προς τον κύριο Ποπόφσκι αγορά το Ντάις, το Ισλαμικό κράτος δηλαδή. Κάποιες από τις υπηρεσίες πληροφοριών μας στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένων και των ρωσικών, πιστεύουν ότι το Ισλαμικό κράτος κατά κάποιο τρόπο προέρχεται από τις ε, ΙΠΑ και από τέτοιου είδους ε, ε, καταστάσεις γιατί βγαίνουν, αποφυλακίζονται κάποια άτομα και Εγώ πιστεύω ότι κανείς δεν μπορούσε να του τροφοδοτεί, κυρίως σε όπλα, δεν υπήρχε συνενοχή κάποιου. Στις υπηρεσίες σας, ε, πιστεύω ότι γνωρίζετε και κάποια άτομα από κάποιες υπηρεσίες πληροφοριών. Ρωτήστε τους κάποια πράγματα και στείλτε μας ένα ενημερωτικό κείμενο. Κάντε το σας παρακαλώ. Δεδομένου ότι τα άτομα τα οποία μου ανέφεραν τέτοιου είδους θέματα είναι σοβαρά, τα γνωρίζω από πολύ καιρό, δεν είναι δικές μου απόψεις. Δεύτερη παρατήρηση. Πώς μπορούμε να διαχειριστούμε αυτή την ανθρωπιστική καταστροφή. Πρώτα απ' όλα, Πρέπει να σας πω ότι την δεκαετία του 80 ήμουν υπεύθυνο της ε, Επιτροπής ε, Ανθρωπιστικής Αποκέντρωσης και βλέπω πόσο συνεχίζει η Αφρική να βρίσκεται σε κακή κατάσταση. Κατάσταση η οποία επιδεινώνεται Όλοι οι κυβερνήσεις είναι πραγματικά με την δική μας συνενοχή ε, κυβερνήσεις που το μόνο που θέλουν να κάνουν είναι να αποκομίσουν ωφέλη. Το λέγω ε, με πλήρη γνώση του θέματος αυτούς. Έτσι δυστυχώς οι Αφρικανοί θέλουν να προς εμάς. Άρα πρέπει να κάνουμε κάτι εμείς για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε την ανάπτυξη αυτής ε, της Υπήρου. Είδαμε τι έγινε στην Λιβύη, στην Συρία, πώς η κατάσταση επιδεινώθηκε και πώς επιδεινώθηκε και το πρόβλημα των μεταναστών, όλων αυτών των ανθρώπων που θέλουν να έρθουν προς εμάς. Κοιτάξτε πώς χειρίζονται με αποτελεσματικό τρόπο κάποιες χώρες τα θέματα αυτά. Η Αυστραλία, η Ελβετία, η Ιαπωνία. Και αντί να κλαψουρίζουμε και να έχουμε λύσεις ε, οι οποίες είναι πραγματικά εφάνταστες αλλά δεν οδηγούν πουθενά, κάντε κάτι το πραγματιστικό και λογικό σε αυτή την Κομισιό. Μήπως δεν θα πρέπει να αναπτύξουμε μία εταιρική σχέση ανάπτυξης για την Αφρική. Με την Κίνα βεβαίως και ασφαλώς και με τη Ρωσία. Με τη Γαλλία που βεβαίως η Γαλλία που γνωρίζει πάρα πολύ καλά την κατάσταση και είναι εγκατεστημένη σε πολλές χώρες δεν μπορεί να κάνει τίποτε από μόνη της. Αλλά βεβαίως μπορεί με νέους εταίρους σημαντικούς να κάνουμε κάτι για να βοηθήσουμε την ανάπτυξη της Αφρικανικής Υπήρου. Αν δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε, το θέμα της μετανάστευσης τώρα μόλις αρχίζει και θα υπάρχουν εκατομμύρια άτομα τα οποία θα θελήσουν τα επόμενα χρόνια και εξαιτία της δημογραφικής πίεσης και της ε, ε, έλλειψης γνώσης του πώς εμείς να την αναπτύξουμε, την Ήπειρο αυτή η οποία έχει και πάρα πολύ μεγάλο φυσικό πλούτο και πλούσιο υπέδαφος, θα δημιουργήσουμε ακόμη περισσότερα προβλήματα. Και αντί για ανάπτυξη θα υπάρχουν σας ευχαριστώ πολύ. Σα ευχαριστώ. ευχαριστώ πολύ για τη συνεισφορά σας. Νομίζω πως εμπλουτίσατε το λεξιλόγιο μας με μια λέξη που δεν έχω ακούσει ποτέ μέχρι τώρα. Που προέρχεται δηλαδή από την Αμερική. Κανένας άλλος δεν ε, το έχει αναφέρει και κανείς δεν έχει, πάρει το, δεν έχει το λόγο, οπότε θα δώσω το λόγο στον κύριο Ποπόφ και για να απαντήσει. Σας ευχαριστώ. Θα είμαι όσο το δυνατόν συντομότερος. Καταρχάς, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει πόλεμο με κανέναν. Όμως, όπως είπε και ο κύριος Φανόρντεν, ο υβριδικός πόλεμος έχει πολλά πρόσωπα και κάποια από τα κράτη-μέλη έχουν ήδη έρθει αντιμέτωπα με κάποιες από αυτές τις μορφές του υβριδικού πολέμου, επιθετική προπαγάνδα για παράδειγμα, ιδιαίτερα σε ορισμένες χώρες στην Ανατολική Ευρώπη. Και αυτό δεν είναι κάτι νέο, υπάρχουν ήδη πάρα πολλές αναφορές στην ρωσική στρατιωτική βιβλιογραφία. Υπάρχει και ένα βιβλίο από το 2007 που αν το διαβάσετε θα καταλάβετε απολύτως τι συμβαίνει στην Ουκρανία αυτή τη στιγμή θα μπορούσαμε να συζητήσουμε αρκετές ώρες για το τι σημαίνει αυτός ο υβριδικός πόλεμος, ε, η επιθετική προπαγάνδα, ε, οικονομικός πόλεμος, άσκηση πίεσης ε, με οικονομικά μέσα κλπ. Τώρα, από το 2003, όταν εγκρίθηκε αρχικά η κοινή στρατηγική, έχουν αλλάξει πάρα πολλά. Καταρχάς τώρα ο κόσμος είναι περισσότερο συνδεδεμένος, όχι μόνο λόγω της ε, τεχνολογικής πρόοδου, αλλά έχουν αλλάξει ε, τα θεμέλια και έχουν τεθεί υπό αμφισβήτηση από πολλά κράτη και από πολλούς ε, άλλους ενδιαφερόμενους φορείς. Είμαστε δηλαδή αντιμέτωποι με, νέου, με, με νέες απειλές, ε, τις ε, κυβερνοεπιθέσεις για παράδειγμα, που τις ονομάζουμε υβριδικές απειλές. Σχετικά τώρα με την προετοιμασία για την κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας που αναφέρατε πολύ, να σας πω ότι η αντιμετώπιση του μεταναστευτικού προβλήματος είναι μόνο μία από τις ε, ενέργειες. Κύριος στόχος είναι να ανασχεθούν οι διακινητές. Και φυσικά ασκείται πίεση και οι χώρες ε, ιδιαίτερα που βρίσκονται στα νότια σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, δέχονται ιδιαίτερα μεγάλη πίεση για να αντιμετωπίσουν αυτές τις ε, μεταναστευτικές ροές. Πιέται επίσης το θέμα της επανεγκατάστασης και μετεγκατάστασης. Ξέρω πως είναι ένα αρκετά ευαίσθητο θέμα και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χθε ενέκρινε κάποιες προτάσεις και τις παρουσίασε μάλιστα και στον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών. Και τώρα αναμένεται να αρχίσει η συζήτηση με τα κράτη-μέλη, τα οποία φυσικά θα πρέπει να εγκρίνουν αυτά τα μέτρα. Και από ό,τι βλέπω αυτό θα γίνει στο τέλος Ιουλίου. Τώρα κύριε Νταντζάν, έχουμε αρκετά ε, μέσα στη διάθεσή μας. Καταρχάς να σας πω ότι εγκρίναμε την εντολή για την αποστολή που αναφέρατε, για τον Ήγηρα, και υποβάλαμε δύο προτάσεις στα κράτη-μέλη. Καταρχάς να επεκταθεί το γεωγραφικό εύρος των επιχειρήσεων και να τους δώσουμε μια εκτελεστική γιατί με αυτόν τον τρόπο οι δικές μας δυνάμεις θα μπορούσαν να συνεργαστούν για την επιτήρηση των συνόρων ε, στον Ήγυρα με τις ε, τοπικές αρχές. Ιδιαίτερα τα σύνορα που βρίσκονται προς την Λιβύη. και να βοηθήσουμε δηλαδή την συνοριοφυλακή εκεί να αντιμετωπίσει αποτελεσματικότερα τις μεταναστευτικές ροές. Με αυτόν τον τρόπο, βοηθώντας εκείνους, βοηθάμε και εμείς τους αυτούς μας φυσικά. Τώρα το πρόγραμμα που δημιουργήθηκε στη Ρώμη σίγουρα δεν είναι όλες οι λεπτομέρειες ε, ολοκληρωσμένες. Σίγουρα πρέπει να συζητήσουμε το τι θα κάνουμε αυτά τα πλοία, πώς θα τα καταστρέψουμε. Και τις επόμενες εβδομάδες αναμένεται να γίνουν συγκεκριμένες προτάσεις γι' αυτό. Τώρα κύριε Βαν Όρντεν, ο στόχος του Συμβουλίου, όπως σας είπα, είναι καταρχάς να δημιουργηθεί μια ισορροπία ανάμεσα στην εφαρμογή και φυσικά να έχουμε την δέσμευση των πολιτικών αρχηγών για τη δημιουργία ενός νέου στρατηγικού πλαισίου. Και επίσης να δούμε πώς θα τονώσουμε και θα ενισχύσουμε τη συνεργασία ανάμεσα στα κράτη-μέλη. Αυτό μπορεί να γίνει για παράδειγμα με διάφορες προπαρασκευαστικές δράσεις και από το Δεκέμβριο του 2013 έχει αλλάξει η διατύπωση. Τώρα διαβάζουμε για πρώτη φορά ότι ε, είμαστε αντιμέτωποι με απειλές στο Νότο και στην Ανατολή. Συζητήσεις με τον ΝΑΤΟ σχετικά με τις επιχειρήσεις στη Μεσόγειο. Να σας πω ότι υπάρχει απόλυτη διαφάνεια πριν την έγκριση της απόφασης πήγα εγώ προσωπικά και ενημέρωσα στο ΝΑΤΟ για τις ε, αποφάσεις εδώ. Πρέπει να συνεχίσουμε να έχουμε καλές σχέσεις με το ΝΑΤΟ, καλή συνεργασία. Ιδιαίτερα για αυτά τα προγράμματα στη Μεσόγειο. Σίγουρα λοιπόν θα συζητηθούν αυτά τα θέματα και πολύ σύντομα. Τώρα, όπως είπατε, πρέπει να γίνει η διοργάνωση από κάτω προς τα πάνω. Και φυσικά γι' αυτό χρειάζεται συνεργασία όλων. Η είπατε εκπρόσωπο συζήτησε το θέμα αυτό όχι μόνο με τους Υπουργούς Άμυνας και Εξωτερικών, αλλά και με τους ε, Υπουργούς Ανάπτυξης την Τρίτη και συμφωνήθηκε ότι χρειάζεται μία ανακατεύθυνση και νέα οργάνωση των συστημάτων σε άλλα μέρη, στην υποσαχάρη Αφρική, στη ζώνη του Σαχέλ, όχι μόνο για να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας, αλλά και για να υπάρχει καλύτερη συνεργασία με τις ε, εκεί κυβερνήσεις που θα οδηγήσει φυσικά στην καλύτερη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών προτού φτάσουν στις ακτές της Λιβύης. Αυτό φυσικά είναι μια δέσμευση μακροπρόθεσμη και δεν μπορεί να γίνει αμέσως, όμως είναι ένας από τους στόχους μας. Εμείς δεν θέλουμε μέσω της ανάπτυξης στρατιωτικών επιχειρήσεων να φέρουμε κάποιο κράτος σε δύσκολη θέση. Θέλουμε πρώτα να είναι καλά ενημερωμένοι όλοι. Γι' αυτό λοιπόν προσπαθούμε να ε, το πράξουμε αυτό, συμμετέχοντας για παράδειγμα σε συνόδους της Αφρικανικής Ένωσης, ενημερώνοντας. Αυτός είναι και ο ρόλος της ΥΠΑ της εκπροσώπου, η οποία τον έχει... Ε, η οποία έχει μεταβεί σε πολλά μέρη και επικοινωνεί με τους ε, αρμόδιους και όσον αφορά τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας να σας πω πως δεν ξέρω πότε θα εγκριθούν υπάρχουν βέβαια κάποιες θετικές εξελίξεις λιγότερες αντιστάσεις στο να δοθεί εντολή στην Ευρωπαϊκή Ένωση όμως δεν έχει ληφθεί ακόμα κάποια απόφαση Και συμφωνώ, οι ίδιοι μετανάστες δεν είναι απειλή. Χρειάζονται προστασία και πρέπει να σεβαστούμε τα δικαιώματά τους. Από την άλλη όμως υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις, μια πρόσφατη περίπτωση σύλληψης ενός υπόπτου, ο οποίος ήταν ύποπτος για τον ε, βομβαρδισμό στην Τινησία. Συνελήφθη στην Ιταλία, πολύ πρόσφατα, και ήταν μέρος ε, μιας ομάδας μεταναστών. Φυσικά αυτό δεν σημαίνει ότι όλοι οι μετανάστες είναι ύποπτοι, όμως πρέπει να έχουμε επαγρύπνηση. Επίσης, στήριξη από τα Ηνωμένα Έθνη. Να σας πω ότι τα Ηνωμένα Έθνη ανέκαθεν ζητούσαν περισσότερη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ε, στρατιωτικέ επιχειρήσει και πιστεύω πως αλλάζουν τα δεδομένα. Δείτε για παράδειγμα τι γίνεται στο Μάλι. Πολλά κρατημέλη, ιδιαίτερα η Σουηδία και οι κάτω χώρε, βρίσκονται στην ε, πρώτη γραμμή και δίνοντας ε, στρατιωτικές ικανότητες και εμπειρογνωμοσύνη. Βρισκόμαστε σε στενή συνεργασία με τα Ηνωμένα Έθνη για τις κοινέ αυτές επιχειρήσεις και ξέρουμε πως αναμένουν από εμάς περισσότερη συμμετοχή. Όπως για παράδειγμα στην περίπτωση του Αφγανιστάν. Όταν αποσύρουν στρατεύματα από εκεί μπορούν να τα στείλουν αλλού. Υπάρχει λοιπόν συνεννόηση. Τώρα, αμυντική βιομηχανία. Δεν θέλω να αναπτύξω το θέμα αυτό πολύ, αλλά να πω πως πράγματι υπάρχουν κάποια γεγονότα. Η αμυντική βιομηχανία έχει ένα αλφαμέγεθος, απασχολεί 800.000 εργαζόμενους στην Ευρώπη και είναι στην πρώτη γραμμή της καινοτομίας. Ας μην το ξεχνάμε αυτό. Η μεγαλύτερες ε, εξελίξεις στην τεχνολογία τα τελευταία 10-20 χρόνια προέρχονται από τον ε, χώρο της αμυντικής ε, βιομηχανίας. Και έρευνα και ανάπτυξη λοιπόν εκεί είναι καλά χρηματοδοτούμενη και πάρα πολύ σημαντική. Τέλος, όπως είπε και ο κύριος Σαφάος, χρειάζεται μία ανάλυση της απειλής. Δεν έχουμε δική μας υπηρεσία πληροφοριών, πράγματι λαμβάνουμε πληροφορίες από τις ε, εκάστοτε εθνικές υπηρεσίες πληροφοριών των κρατών μελών. Και τις χρησιμοποιούμε για να μπορέσουμε να λάβουμε τις ε, σωστές αποφάσεις. Ιδιαίτερα, για παράδειγμα, στην περίπτωση του Ισλαμικού κράτους. Και να πω κάτι για την πολιτική ασφάλειας και Άμυνα Μάλλον τον Νοέμβριο, όπως επιβεβαιώθηκε στην έκτακτη συνεδρία του Συμβουλίου τον Απρίλιο, θα γίνει μια σύνοδος που, στην οποία θα συμμετέχουν πολλές αφρικανικές χώρες, στη Μάλτα, ακριβώς για να συζητηθεί το θέμα της εμαζικής μετανάστευσης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Ποπόφσκι για τις επεξηγήσεις σας και για τις απαντήσεις σας. Βλέπω ότι ο κύριος Βεράσκη θέλει να μιλήσει. Θα, θα κλείσουμε την ε, συζήτηση, αλλά ε, γρήγορα μπορείτε να πείτε κάτι αν θέλετε. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κοιτάξτε, Παρακολούθησα με προσοχή τη συζήτηση και πρέπει να πω ότι με προβληματίζει η δέσμευση η οποία όμως ε, δεν φαίνεται να μπορεί να φέρει πολύ καλά αποτελέσματα. Κατά την άποψή μου, ο ευρυδικός πόλεμος χρήζει υβριδικής απαντήσεως. Ε, οι εχθροί της ειρήνης, των δικαιωμάτων των ανθρώπων ε, και της δικαιοσύνης και της δημοκρατίας χρησιμοποιούν και τον πραγματικό χώρο και τον κυβερνοχώρο. Ε, εμείς όμως αντιμετωπίζουμε αυτές τις υβριδικές ε, απειλές με, τα, με τον παλιό τρόπο. Λες και θέλουμε τώρα να προχωρήσουμε στο μέλλον οδηγώντας μία τράμπαντ. Ένα αυτοκίνητο πολύ παλιού μοντέλου. Αυτός ο υβριδικός πόλεμος πρέπει να ε, ε, χτυπηθεί με, νέα, ε, με νέους τρόπους, νέα εργαλεία, με μια υβριδική απάντηση, ανταπόκριση εν πάση περιπτώσει. Υπάρχουν οπωσδήποτε κάποια στοιχεία τα οποία σιγά σιγά σχεδιάζονται αλλά δεν υπάρχει ένα συνολικό ε, πρόγραμμα. Δεν θα έχουμε ποτέ ε, στρατό ευρωπαϊκό, αλλά θα πρέπει η διαφορετική μας στρατή στην Ευρώπη, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να εξειδικευτούν περισσότερο και να έχουν την δυνατότητα να δώσουν αυτήν την ε, υβριδική απάντηση στον υβριδικό πόλεμο. Ένα τελευταίο. Τέλη Μαΐου βρισκόμαστε πλέον και γνωρίζουμε Γνωρίζουμε, λέω, ποιες είναι οι ε, χρηματοδοτικές ικανότητες που μπορούμε να έχουμε. Τις γνωρίζουμε αυτές ή τίποτα. Ευχαριστώ πολύ για τα σχόλιά σας, ε, κύριε Ζρογεύσκη. Νομίζω ότι θα έχουμε ούτως ή άλλως περισσότερες ευκαιρίες να δώσουμε τον ε, λόγο στους κυρίους στο πάνελ για να απαντήσουν. Τώρα θα ήθελα να καλωσορίσω τον επόμενο καλεσμένο μας, τον κύριο Μάρκους Κορνάρο, ο οποίος ε, είναι αναπληρωτής γενικός διευθυντής ε, για, την, ε, για τον γεωγραφικό συντονισμό της Γενικής Διεύθυνσης ΔΕΒΚΟ. Ε, υπάρχει μια πρωτοβουλία την οποία γνωρίζουμε, την ονομάζουμε Train and Equip. Δεν πρόκειται για νέα πρωτοβουλία. Θυμίζω ότι πολλά χρόνια πριν ε, οι επικεφαλείς μας στο Αφγανιστάν χρησιμοποιούσαν την μέθοδο αυτή μαζί με τους Αμερικανούς στρατιώτες εκπαίδευαν και τους Αφγανούς στρατιώτες αλλά ε, πριν τους μάθουν στρατιωτικό βηματισμό έπρεπε να τους δώσουν παπούτσια γιατί δεν είχαν καν ε, παπούτσια αυτό ήταν, αυτό ήταν το πνεύμα ποιο είναι το όριο του εξοπλισμού που παρέχεται σε άλλους στρατούς. Ξεκινάμε από παπούτσια, ε, φτάνουμε σε ε, αλεξίσφαιρα γυλαίκα, ε, μιλάμε και για κάτι άλλο. Θα μπορούσατε ε, ε, αγαπητοί μου να μας απαντήσετε σε αυτές τις ερωτήσεις που είναι οι ερωτήσεις μου. Ε, βέβαια πρώτα θα κάνετε τις αρχικές σας τοποθετήσεις. Θα δώσω πρώτα το λόγο για τις παρουσιάσεις και μετά τα ερωτήσεις. Ο κ. Ποπόφσκι. Κοιτάξτε, εγώ μεγάλωσα κοντά στα τσεχικά σύνορα, ξέρω πολύ καλά. Καταλαβαίνω κιόλα τι λέτε. Πρώτα μία απάντηση στον κύριο Στραγεύσκη όσον αφορά το, την υβριδική ανταπόκριση στον υβριδικό πόλεμο. Συμφωνώ απολύτω και είναι ένας εκ των λόγων για τον οποίο η ύπατη αντιπρόσωπος ε, θα παρουσιάσει ε, μία έκθεση τον Ιούνιο ακριβώς για αυτό το θέμα. Επίσης να απαντήσω στην ερώτηση του κυρίου Ντονζόν όσον αφορά την χρηματοδότηση της πολιτικής ασφάλειας και άμυνας. Πρέπει να είμαι ειλικρινής, γιατί έτσι το έθεσε και στα κράτη-μέλη, η εκπρόσωπος. Ε, με το πρόγραμμα Αθήνα καταφέραμε να κρατήσουμε το status quo, δεν, δεν πήγαμε παραπέρα. Νομίζω ότι με τον τρόπο αυτό θα μπορέσουμε να χρηματοδοτήσουμε επαρκώς ή τέλο πάντων να έχουμε μια ικανή χρηματοδότηση των ε, μη στρατιωτικών ε, ε, στοιχείων της πολιτικής ασφάλειας και άμυνας. Τώρα δεν ξέρω εάν θα έχουμε συγκεκριμένο ε, ε, αριθμητικό στοιχείο, συγκεκριμένο ποσό για το ξεκίνημα των επιχειρήσεων. Τέλος πάντων, όσον αφορά την equip, Train and Equip, τώρα όμως η επίσημη ονομασία είναι Capacity Building in Support of Development. Αυτό αναφέρεται και στο κοινό ανακοινωθέν της Υπηρεσίας Κριτικής Δράσης και της Κομισιόν. Ε, βάσει αυτών των στοιχείων που είχαμε θέλαμε να υπάρχει ενότητα στόχου όταν βρισκόμαστε σε τρίτες χώρες. Πρόκειται για μία έννοια, για ένα κόνσεπτ το οποίο θα θέλαμε ε, να υποβάλουμε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το οποίο άλλωστε είχε αιτηθεί ενός μια τέτοιας σκέψης. Βασιζόμαστε στην επιχειρησιακή μας επιτόπου και επί του ε, ε, πραγματογνωμοσύνη. Έχουμε αρκετή πραγματογνωμοσύνη σε αφορά τα θέματα αυτά, αλλά υπάρχουν και όρια. Ας πούμε, εκπαιδεύσαμε πολλούς στρατιώτες στο Μαλί και στη Σομαλία, ε, ίσως 7-8 χιλιάδες μέχρι το τέλος του έτους, αλλά δεν μπορούμε ή τέλο πάντων έχουμε σημαντικούς περιορισμούς ε, να τους δώσουμε τον εξοπλισμό που χρειάζονται. Είτε πρόκειται για όπλα, ε, είτε πρόκειται και για πολύ απλά πράγματα τα οποία χρειάζεσαι έτσι ώστε ε, να μπορέσει να κάνεις τη δουλειά σου, δηλαδή οχήματα, υλικό επικοινωνία κτλ. Πρέπει λοιπόν να προσαρμόσουμε την πολιτική μας ε, έτσι ώστε να είμαστε σε θέση ε, να βοηθήσουμε λαμβάνοντας υπόψη τους νομικούς και λοιπούς περιορισμούς. Να δούμε πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας ή άλλα εργαλεία. Η εμπειρία μας συνδέεται κυρίως με αυτά που είπα προηγουμένως Μαλή ε, και Σομαλία. Τώρα θα πάμε και σε άλλες χώρες με την ίδια αρχιτεκτονική. Πρώτα απ' όλα βλέπουμε το υφιστάμενο ε, ρυθμιστικό πλαίσιο το οποίο αναφέρεται άλλωστε και στις συνθήκες Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης ε, και βλέπουμε και τους κανόνες της, του ΑΣΕΝΤΑΚ και όλες τις άλλες σχετικές, όλα τα άλλα σχετικά εργαλεία, κυρίως το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης. Ε, το σημαντικό είναι να υπάρχει συνοχή ε, στην ε, δράση μας και αυτό εξαρτάται εν μέρει και από τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα ήδη υφιστάμενα εργαλεία. Τώρα, ποιες είναι οι κατηγορίες της εργασίας, των εργασιών που έχουμε μπροστά μας. Πρώτα απ' όλα πρέπει να βελτιώσουμε το συντονισμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τα κράτη-μέλη και άλλους εμπλεκόμενους, οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι Ηνωμένα Έθνη κυρίως. Ε, θα πρέπει να μελετήσουμε ε, τα πράγματα έτσι ώστε να ε, παράσχουμε ένα καλό πλαίσιο για παρέμβαση και τέλος να, βρούμε, να δούμε τα χρηματοδοτικά και ρυθμιστικά μέτρα. Όσον αφορά το τελευταίο, πρέπει να μελετήσουμε την πρακτική εφαρμοσιμότητα τριών δράσεων. Πρώτα απ' όλα η προσαρμογή της Africa Peace Facility. Είναι ένα εργαλείο το οποίο γνωρίζετε, ξεκίνησε το 5 αν δεν κάνω λάθος και Έχουμε ξοδέψει 1,2 ε, δις ε, ευρώ από τη στιγμή της σύλληψης και ε, χρήσης αυτού του εργαλείου, αλλά υπάρχουν περιορισμοί και θέλουμε να μελετήσουμε γενικότερα το θέμα και από τη στιγμή που ε, ε, το Αναπτυξιακό Ταμείο είναι αυτό το οποίο χρηματοδοτεί ε, το εργαλείο που ανέφερα πρέπει να το δούμε. Μετά θα πρέπει να δούμε την διασύνδεση ανάμεσα στη χρηματοδότηση και την διαδικασία ειρήνευσης και διατήρησης της ειρήνης. Θα πρέπει να δούμε αν θα έχουμε ένα εργαλείο ή πολλά. Τρίτον, η τρίτη ιδέα η οποία είναι νέα είναι ε, ε, η δημιουργία ενός νέου ε, αποκλειστικής χρήσης εργαλείου οικοδόμησης ικανότητας. Ε, ε, με τον τρόπο αυτό θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε συνολικά όλα αυτά τα ζητήματα τα οποία σας ανέφερα προηγουμένως. Τα κράτη-μέλη επίσης καλούνται ε, να δουν το ενδεχόμενο διεύρυνση του μηχανισμού ΤΙΝΑ έτσι ώστε να ληφθούν νέες ε, διευθετήσεις ε, ε, και βέβαια υπό τον άμεσο έλεγχο Κομισιόν και Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης. Πρέπει να ξεκινήσουμε την δράση. Αυτή είναι άλλωστε και η αρχή της αντίληψης που έχουμε. Να ξεκινήσουμε από το Μαλί, από την Σομαλία, να ε, έχουμε και την ε, ε, και να έχουμε και την γενικότερη έποψη. Κοιτάξτε, δεν είναι αποκλειστική η ενασχόλησή μας με την Αφρική, απλώς είναι αφρικοκεντρική. Από τη στιγμή που θα... Ε, αυτό που θέλουμε εμείς είναι ε, να μην, ε, να μην περιορίσουμε την γεωγραφική εμβέλεια του εργαλείου και αυτό θέλουμε να το καταστήσουμε σαφές στις χώρες μέλη. Και βεβαίως εδώ μας βοηθούν και η Γενική Διεύθυνση ΤΕΒΚΟ και άλλες υπηρεσίες. Εδώ μιλάμε για βασικά πράγματα, νομική βάση, περιορισμοί που πρέπει να αντιμετωπιστούν, αλλά νομίζω ότι πάντως τα πρώτα στοιχεία είναι αρκετά ενθαρρυντικά. Είναι πολύ ικανοποιητική η κοινή μα εργασία. Περιμένουμε τώρα να δούμε τι λόγο θα έχουν οι υπουργοί, πώ θα αντιμετωπίσουν το θέμα. Θα δούμε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και προσδοκούμε να μας δώσει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και κάποιο περιθώριο ελιγμών έτσι ώστε να μπορέσουμε ε, να κινηθούμε στην πράξη. Πιστεύω ότι υπάρχει μεγάλος βαθμός απέτησης έτσι ώστε να υπάρξει μεγαλύτερη οικοδόμηση ικανοτήτων ε, και βεβαίως αυτό θα το δούμε και σε συνδυασμό με την αντιμετώπιση ε, των προβλημάτων των μεταναστευτικών ροών στη ρίζα τους. Ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ κύριε Παπόφσκι. Κύριε Κορνάρο, σας δίνω το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ. Αγαπητά μέλη, με χαρά μου να ακολουθήσω τον κύριο Ποπόφσκι Το θέμα αυτό είναι ένα θέμα που μας έφερε πολύ κοντά τους τελευταίους μήνες. Υπάρχει έλλειψη διακυβέρνησης, αυξημένη φτώχεια και όλα αυτά έχουν πολύ έντονες συνέπειες στην ασφάλεια. Αυτό είναι μια διαπίστωση στην οποία έχουμε καταλήξει χρειάζεται να αντιμετωπιστούν αυτές οι προκλήσεις από όλους και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από τους ε, τοπικούς παράγοντες. Για να γίνει αυτό χρειάζεται εμείς να παρέχουμε ολοκληρωμένη στήριξη έτσι ώστε οι εταίροι μας να μπορέσουν να δημιουργήσουν τις δικές τους ε, ικανότητες σχετικά με την ασφάλεια. και δημιουργία ικανοτήτων δηλαδή, όχι όμως μόνο για την ασφάλεια, αλλά και για την ε, κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη. Πιστεύω πως η ανακοίνωση την οποία εγκρίναμε τον Απρίλιο το αναφέρει ρητά και το θέτει ως κύρια προτεραιότητα. Εντοπίζονται κάποια κενά και κάποιες ελλείψεις στην ε, ανταπόκριση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επίσης προτείνονται κάποιες λύσεις, τις οποίες θα σας ε, αναφέρω διεξοδικότερα αργότερα. Σε γενικές γραμμό, γραμμές να σας πω ότι υπό το υφιστάμενο πλαίσιο χρειάζεται βελτίωση στην προσέγγιση της Ευρώπης στην ασφάλεια και την ανάπτυξη και επίσης ανάπτυξη ενός ε, συνεκτικού πλαισίου για τον έλεγχο και παρακολούθηση και την διαχείριση των κινδύνων. Αυτές είναι οι δύο κύριες ε, κατευθύνσεις τις οποίες έχουμε. Και όπως τόνισε και ο κύριος ε, Ποπόσκι, προσπαθούμε να εξετάσουμε και το πόσο εφικτές είναι αυτές οι νέες ε, προτάσεις. Θέλουμε λοιπόν να προωθήσουμε μια πιο ισορροπημένη, πιο συνεκτική προσέγγιση της, στην αντίδραση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία θα συμφωνεί και θα συνάδει με τις ε, εθνικές πρακτικές, έτσι ώστε να είναι και πιο αποτελεσματική. Τα συμπεράσματα του Συμβουλίου του Μαΐου για την κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνα είναι αρκετά φιλόδοξα και αναμένουμε το Συμβούλιο του Ιουνίου να δώσει την κατάλληλη πολιτική καθοδήγηση για την υλοποίησή τους. Και θα ήθελα να επαναλάβω και εγώ ότι Χωρίς ανάπτυξη δεν υπάρχει ασφάλεια και αντίστροφα, χωρίς ασφάλεια δεν υπάρχει ανάπτυξη. Πρέπει να το έχουμε υπόψη αυτό. Γι' αυτό λοιπόν ε, θα σταματήσω εδώ και θα ήθελα να ευχαριστήσω εσάς κύριε Πρόεδρε που μας καλέσατε εδώ για να ενημερώσουμε την Επιτροπή σας διότι μην ξεχνάμε ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι πάρα πολύ σημαντικός έχει νομοθετικές αρμοδιότητες και αυτές πρέπει να τις χρησιμοποιήσει όσο το δυνατό περισσότερο και στο μέλος Επίσης θα ήθελα να πω πως εμείς θα επιθυμούσαμε και η Επιτροπή Ανάπτυξης να συμμετέχει στις διαβουλεύσεις που κάνουμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πιστεύω πως και ως μέλος της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, η συμμετοχή της δικής Επιτροπής ε, Ανάπτυξης είναι πάρα πολύ σημαντική. Τώρα, όπως είπα, θα αναπτυχθώ σε αυτά που είπατε αργότερα. Όμως θα ήθελα να σταθώ σε δύο θέματα. Καταρχάς, η ανακοίνωση δηλώνει σαφέστατα ότι θα κινηθεί μόνο εντός των νομικών ορίων που έχει. Έπειτα υπάρχουν συγκεκριμένες αναφορές σχετικά με το ε, τι θεωρείται πραγματική ανάπτυξη. Ακολουθούνται τα πρότυπα του ΩΣΑ και οι κατευθυντήριες του γραμμές. Τι σημαίνει αυτό. Με πολύ λίγες εξαιρέσεις δηλαδή οτιδήποτε συνδέεται με στρατιωτικές επιχειρήσεις δεν ε, γίνεται αποδεκτό ως ε, ανάπτυξη. Καλωσορίζω κλείνοντας ε, όλη την προσπάθειά σας και την πρόσκλησή σας και είμαι ανοιχτή σε ερωτήσεις. Σας ευχαριστούμε και εμείς κύριε Κορνάρο. Θα αρχίσουμε τώρα την ανταλλαγή απόψεων. Έχετε το λόγο κύριε Τάνσο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Η Πέμπτη του πρωί είναι μία πολύπλοκη μέρα. Για να συζητήσουμε όμως κατά την άποψή μου μία τόσο σημαντική πρωτοβουλία, πολλές φορές ε, ήδη το συζητήσαμε, αλλά έχουμε πολύ λίγες φορές τόσο συγκεκριμένα και σημαντικά θέματα τα οποία περιμένουμε από το Συμβούλιο των Ιούνιων. Τώρα, Όσον αφορά το πρόβλημα αυτό, train and equip, πρέπει να πω ότι είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα προς ώστε στη δράση μας να δώσουμε αποτελεσματικότητα σε θέματα ασφάλειας και ανάπτυξης. Είναι ένα πρόγραμμα για το οποίο μιλούμε εδώ και πάρα πολύ καιρό. Και όπως είπατε, οι ελλείψεις εντοπίστηκαν εδώ και πάρα πολύ καιρό. Υπενθυμίσατε ότι η υποεπιτροπή ε, πήρε μέρος σε διάφορες στρατιωτικού τύπου και μη αποστολές στις χώρες αυτές και πάντα ακούγαμε τα ίδια σχόλια. Δηλαδή, να μας συμβουλεύετε, να μας ενημερώνετε, καλό είναι, πλην όμως αν δεν έχουμε τον κατάλληλο εξοπλισμό δεν μπορούμε να ενεργήσουμε αποτελεσματικά. Και όταν μιλούμε για εξοπλισμό δεν μιλούμε για τάγκς, δεν μιλούμε για μηχητικά αεροπλάνα στο η Νέστορ, ΙΚΑΠ για το κέρας της Αφρικής μιλούμε για εξοπλισμό ασφάλειας για υπολογιστές πολλές φορές για εργαστήρια για την επιστημονική ε, αστυνομία εξοπλισμό ο οποίος δεν είναι καθόλου δαπανηρό σε σχέση με τα χρήματα που δαπανούμε αλλού. Είναι λοιπόν πρωταρχική σημασία να παρακολουθήσουμε αυτή την κατάσταση και να δώσουμε συνέχεια σε αυτό που κάνουμε. Τώρα, η θεωρία ωραία. Αλλά στην πράξη, όπως ξέρουμε και λέμε, ο διάβολος βρίσκεται στις λεπτομέρειες. Ας το προσέξουμε αυτό. Είπατε κύριε Ποπόφσκι ότι μελετάτε πολλά επιμέρους θέματα. Εγώ πρέπει να ομολογήσω το εξής. Η δημιουργία ενός ειδικού ε, κονδυλίου για την υλοποίηση αυτού του στόχου νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντική. Και επανέρχομαι σε αυτό που είπατε που είναι τόσο σημαντικό. Το είπατε και δύο. Ο συντονισμός, η συνοχή. Δεν είναι ότι δεν γίνεται τίποτα στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το Train and Equip. Πάρα πολλά όμως κατακαιρματισμένες προσπάθειες Χωρί συντονισμό μεταξύ του, Πράγμα το οποίο δημιουργεί και τρομερή σύγχυση στους εταίρους μα. Ποιο κάνει τι, σε ποιον πρέπει να απευθυνθώ, η Επιτροπή, το Συμβούλιο, τα κράτη-μέλη. Ακούστε, πρόκειται πραγματικά για τρόπο δράσης που και εγώ πολλές φορές δεν καταλαβαίνω. Πηγαίνει κανείς ε, στην ε, Αφρική, στο κέντρο της Αφρικής όλοι μας λένε είναι comprehensive crowd, σφαιρική προσέγγιση. Αλλά δεν ξέρει κανείς ούτε ποιος κάνει τίποτα, ούτε ποιος ηγείται κανένας προγράμματος. Ούτε και εγώ καταλαβαίνω. Καταλαβαίνετε λοιπόν οι δικαιούχοι, τα αφρικανικά κράτη, αυτού του οποίου απευθύνονται αυτά τα προγράμματα τι κάνουν. Και ο Ευρωπαίος φορολογούμενος χρηματοδοτεί αυτές τις δράσεις και επίσης δεν καταλαβαίνει τίποτε. Διαθέτουμε κονδύλια, δεν ξέρει ποτέ κανένα τι κάνουμε. Πρέπει λοιπόν να ενεργήσουμε ορθολογικά. Μιλάτε για συνεκτικότητα και συντονισμό. Εμένα δεν μου αρέσει η έλλειψη, το θέμα του συντονισμού. Τι σημαίνει όμως συντονισμός εδώ. Έχουμε δύο δομές που ε, η καθεμία κάνει κάτι και θα δημιουργήσουμε μία τρίτη δομή για να συντονίσει αυτό που κάνει οι άλλες δύο. Τέλος πάντων, είναι λίγο ε, επιγραμματικά αυτά που λέω και σαν καρικατούρα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, δεν χρειάζεται να δημιουργήσουμε ένα νέο χρηματοδοτικό μέσο. Νομίζω ότι έχουμε πάρα πολλά είδη τα οποία θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε σωστά. Μην δημιουργούμε λοιπόν επαχθείς γραφειοκρατικές δομές περαιτέρω. Δεν θα διευκολύνουμε τα πράγματα. Ελπίζω ότι θα μπορέσετε με ευελιξία και λογική να χειριστείτε το θέμα αυτό, δεδομένου ότι υπάρχει επίγουσα ανάγκη. Χαιρετίζω το γεγονός ότι και στην ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στον ε, ε συμμεριζόμαστε τις ίδιες ιδέες. Ελπίζω λοιπόν ότι θα μπορέσουμε με λογική να καταλήξουμε σε κάτι το οποίο θα είναι αποτελεσματικό. Σας ευχαριστούμε κύριε Ντονζό. Η κυρία Σεμπάγιος. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Συμφωνώ απολύτως με τον κύριο Κορνάρο, ε, με την έννοια δηλαδή ότι δεν υπάρχει ασφάλεια ε, χωρίς ανάπτυξη ή ανάπτυξη χωρίς ασφάλεια. Επομένως θα πρέπει οπωσδήποτε ε, να δουλέψουμε για τα θέματα της καλής ε, διακυβέρνησης και να βοηθήσουμε και στις αναπτυσσόμενες χώρες, αλλά θα πρέπει να κάνουμε ένα καλό παιχνίδι ισορροπιών. Θα πρέπει να καταλάβουμε πρώτα απ' όλα ποια είναι, τι είναι η βοήθεια ε, και να προσπαθήσουμε να ξεχωρίσουμε τα στρατιωτικά από τα μη στρατιωτικά. Λείπει, λείπει ο έλεγχος και η λογοδοσία και ο κοινοβουλευτικός έλεγχος. Πώς θα διαρθρωθούν όλα αυτά τα πράγματα. Τι γίνεται με την διαφάνεια, με την, με την καλή διακυβέρνηση είναι σημαντικό με κάποιο τρόπο να διασφαλιστεί η ε, αλλαγή. Εμείς σαν πράσινοι θέλουμε να δούμε αλλαγή. Θέλουμε να γίνει περισσότερος λόγος ε, για κατάρτιση, για χρηματοδότηση ε, και για εξοπλισμό όσον αφορά τις δυνάμεις ασφαλείας σε αυτές τις εμπλεκόμενες χώρες. Ε, αυτό το ντάκαμπολ επίσης ε, ε, κοιτάξτε, είναι εδώ και πολλά χρόνια ε, βλέπουμε ότι πολλές χώρες προσπαθούν να κερδίσουν από τον ε, στρατιωτικό τομέα όσον αφορά τη, τον κανονισμό DAC. τι σημαίνει δηλαδή να πρέπει να μπορεί να ανάγεται στον κανονισμό DAC. Ε, αυτό που μπορώ να πω εγώ είναι ότι ε, πολύ λιγότερο γίνεται αυτή η αναγωγή στο ΤΑΚ ε, στις περισσότερες χώρες και από την άλλη πλευρά το να βγάζουμε απ' έξω οτιδήποτε δεν, δεν ονομάζουμε και δεν ορίζουμε ως ντάκαμπολ εντός εισαγωγικών δεν είναι και σωστό. έπτα ε, αναφέρεται, επιπλέον γράφεται εδώ, επιπλέον περιορισμοί ε, τι σημαίνει περισσότεροι ε, περιορισμοί. Αυτό νομίζω ότι είναι επικίνδυνο και σε σχέση με τον κανονισμό DAC. Επίσης στη σελίδα 11, στη σελίδα 11 λέτε ε, ότι θα πρέπει ε, η ειρήνη και ε, να να ληφθούν υπόψη λαμβάνοντας υπόψη και τα όσα αναφέρονται και στη σελίδα 9 και ε, τους περιορισμούς βλέπετε και στη σελίδα 9 και στη σελίδα 11 έχουμε πρόβλημα όσον αφορά την έννοια των περιορισμών υπάρχουν πράγματα τα οποία ενδεχομένως δεν μπορούν να γίνουν τώρα αλλά θα γίνουν στο μέλλον Děkuji. Eh, Αν μου επιτρέπετε, θα ήθελα και εγώ να σας κάνω μια ερώτηση που έχει σχέση με την πρωτοβουλία Train and Equip. Εκπαιδεύω και εξοπλίζω. Και μιλούμε κυρίως για την Αφρική. Η πρωτοβουλία αυτή θα μπορούσε να διευρυνθεί και να εφαρμοστεί και σε άλλες χώρες όπως Φερρυπίν στην Ουκρανία. Εγώ πρόσφατα επισκέφθηκα την Ντόμπας και συνάντησα εθελοντές στρατιώτες και όταν είδα τις μπότες που φορούσανε τι να πω πέδιλα μάλλον φορούσαν μερικοί αντί για μπότες στρατιωτικές αυτές ε, λοιπόν ε, ε, οι στρατιώτες που δεν είναι μέρος του επίσημου στρατού, αυτά τα εθελοντικά στρατεύματα δεν έχουν κανένα εξοπλισμό αλλά προστατεύουν κάποια μέρη και διαρωτώμε θα μπορούσαμε στα πλαίσια αυτής ε, της πρωτοβουλίας να συμπεριλάβουμε και την Ουκρανία επειδή δεν υπάρχουν άλλες ε, ερωτήσεις Σα δίνω το λόγο και αποφασίστε εσεί ποιο θα αρχίσει πρώτος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα, μια γενική παρατήρηση. Όλα αυτά αποτελούν μέρο γενικότερη ιδέα τη διακυβέρνηση. Δεν μπορούμε να είμαστε σοβαροί αν θέλουμε να κάνουμε σωστή διακυβέρνηση στην Αφρική χωρί το θέμα τη ασφάλεια να το χειριστούμε. Διαφορετικά τι κάνουμε. Μπορούμε να κάνουμε δικά δίκτυα και σχολεία αν δεν υπάρχει όμως ε, σωστή αστυνομία και στρατός που δεν έχει διαφθαρεί δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα για την ανάπτυξη της χώρας. Και βεβαίως η οποιαδήποτε σημαντική και σοβαρή πρωτοβουλία και θέλουμε να είμαστε σοβαροί γνωρίζοντας συγχρόνως ποιοι είναι οι περιορισμοί ενέχουν και αυτό το στοιχείο της ασφάλειας και ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Είπε κάτι ο Μάρκος για την ε, συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνο όταν θα μπορέσουμε να έχουμε τη σωστή ε, νομική βάση και εσείς συναποφασίζετε ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε σωστά. Τώρα αν θα είναι μέρος της αναθεώρησης ή στα πλαίσια μίας, του, της ε, επόμενης ε, δημοσιονομική, δημοσιονομικού προγραμματισμού που θα γίνουν για τα επόμενα χρόνια θα το δούμε. Το 2005-2006 στην Επιτροπή είχε δημιουργηθεί το μέσον αυτό για την σταθερότητα όπως το ονομάζουμε σήμερα και νομίζω ότι μπορούμε τα μέσα που έχουμε να κάνουμε κάποια πράγματα αλλά ίσως όχι μέχρι εκεί που θα θέλαμε. Σας κάνουμε έκκληση. Εάν θέλετε και σας θέλουμε μαζί μας, κάντε κάτι κι εσείς από νομαστικής πλευρά για να προχωρήσουμε πιο αποτελεσματικά. Δεν ε, θέλω ε, να τονίσω το σκέλος το στρατιωτικό στα πλαίσια της ανάπτυξης. Αλλά θα σας πω το εξή. Και άλλοι είναι αυτοί οι οποίοι ε, ασχολούνται με τα θέματα της αναπτυξιακής βοήθειας, όπως το Ηνωμένο Έθνη. Η πρόθεσή τους δεν είναι να δούνε ποια είναι ε, τα αποτελέσματα αποκλείοντας κάποιους. Εάν οι στρατιωτικοί μπορούν επίσης να κάνουν κάτι στα πλαίσια τη συνεργασία για να υπάρξει ανάπτυξη, είναι κάτι το οποίο μπορούμε να το προβλέψουμε. Με τα μέλη της Ντάκα αυτής της Επιτροπής για την Αναπτυξιακή Βοήθεια και από μεριάς Ευρώπης έχουμε με τους υπόλοιπους πολύ καλή συνεργασία. Και ελπίζουμε ότι μέχρι το τέλος του έτους θα μπορέσουμε κάποιους κανόνες στα πλαίσια ε, της συνεργασίας να τους επικαιροποιήσουμε για να προχωρήσουμε. Δεν είναι μόνο μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση εκεί, είναι και η Νορβηγία φέρει μεταξύ άλλων. Τώρα, οι ορισμοί και οι γραμμές πλεύση που είχαμε καθορίσει πριν από 10 χρόνια δεν ισχύουν ε, ενδεχομένως σήμερα διότι η έχουν αλλάξει πολλά πράγματα. Θα αναφέρω κάτι το οποίο αφορούσε τον ε, ε, στρατό στο Κονγκό, κάποια χρήματα τα οποία ε, αφορούσαν τους στρατιώτες, αλλά άλλαξαν τα πράγματα. Δεν μπορούμε να ότι αυτό μπορεί να θεωρηθεί ως ενίσχυση ότι είναι, γίνεται στα πλαίσια της Επιτροπής Αναπτυξιακής Βοήθειας. Νομίζω πρέπει να κάνουμε μία συζήτηση πολύ σοβαρή γραμμή προς γραμμή να δούμε τα κονδύλια του προβλήματος που δίνονται και για ποιο σκοπό για να προχωρήσουμε. Με πιο σύγχρονο τρόπο αν θέλετε. Υπάρχουν δύο-τρεις σημαντικές ιδέες τις οποίες θα προχωρήσουμε. Θα δούμε και από νομικής πλευράς ε, οι ορισμοί πώς ε, εφαρμόζονται σήμερα. Όσον αφορά ε, τα μέσα αυτά που αφορούν την ανάπτυξη και τις υποδομές για την Αφρική θα τα εξετάσουμε. Πιστεύω ότι στα πλαίσια των μέσων για τη στήριξη της ειρήνης της Αφρικής μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και παραδείγματα ή μέσα που χρησιμοποιήσαμε για τα Βαλκάνια, για κάποιες χώρες, για τη Μολδαβία, αλλά θα πρέπει να έχουμε μια σφαιρική προσέγγιση και να δούμε ότι χρησιμοποιήθηκε αλλού, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και εκεί επωφελώς. Ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα, για να απαντήσω στον κύριο Νταζό, σας ευχαριστώ για την ανάλυση σας και διότι ε, αναφέρατε το πόσο πολιτικά σημαντικό είναι το θέμα αυτό και η ανταπόκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πρέπει να είναι πολιτική επίσης. Μπορώ να σας διαβεβαιώσω για το εξής. Δεν φοβούμε ότι θα χαθούμε σε γραφειοκρατικές ατέρμονες συζητήσεις. Όλοι συνειδητοποιούμε το ότι θα πρέπει πρώτα απ' όλα σε πολιτικό επίπεδο να σκιαγραφίσουμε τον δρόμο που θέλουμε να ακολουθήσουμε και τα μέτρα που θέλουμε να λάβουμε εμείς στην Ευρώπη. Βεβαίως λαμβάνοντας υπόψη τη νομική βάση για να λύσουμε αυτά τα προβλήματα που προαναφέρατε και ελπίζω ότι στο Συμβούλιο τον Ιούνιο και στις ε, μετέπειτα συζητήσεις θα διευκρινιστούν όλα αυτά τα θέματα. Ε, Τώρα, την ε, ανακοίνωση όσον αφορά το πολιτικό σκέλος. Γίνεται λόγος για την αξιολόγηση κινδύνου. Εσείς μιλήσατε για την ε, Ουκρανία. Εγώ ε, παρακολούθησα εκ του σύνεγγυς τα γεγονότα στις πλατείας Τιενανμέν. Το ερώτημα είναι μέσα που χρηματοδοτήσαμε για να βοηθήσουμε την αστυνομία χρησιμοποιήθηκαν τότε για να πολεμήσει τους ε, αντίθετους προς τις ιδέες αυτές η αστυνομία. Υπάρχουν ακόμη ερωτηματικά για το θέμα αυτό. Πλην όμως θα πρέπει να σκεφτούμε τι έγινε με τον εξοπλισμό που έστειλε στο Μαλή η Γαλλία, που χρησιμοποιήθηκε κάποια στιγμή από κάποιους εξεγερμένους. Τώρα, εμείς, στην Ευρώπη, από πολιτικές πλευράς, το Κοινοβούλιο, προς τους πολίτες, τι έχουμε να πούμε. Ίσως κάποια εξοπλισμούς που στείλαμε και χρηματοδοτήσαμε βρίσκονται στην κακιά πλευρά σήμερα. Θα πρέπει όμως να, και το συνειδητοποιούμε αυτό, να προσέξουμε πάρα πολύ το πώς θα πρέπει να δούμε πώς έχει η εκεί πραγματικότητα για να βρούμε τις κατάλληλες και πιο αποτελεσματικές λύσεις. Και τώρα ακόμη κάτι το οποίο είναι πιο δύσκολο αλλά από το train and equip είναι το capacity building. Η δημιουργία ικανοτήτων υποδομών δηλαδή που μπορούμε να βοηθήσουμε να αναπτυχθούν και να δούμε σε ποια δυναμική, με ποια δυναμική και με ποιες προοπτικές εργαζόμαστε ώστε εμείς στα πλαίσια της ανάπτυξης να εξασφαλίζουμε ότι ό,τι κάνουμε ε, γίνεται σωστά αποδεκτό από τους εταίρους μας building του... Um, uh, uh, Τέλος πάντων θα πρέπει ότι κάνουμε να είμαστε σίγουροι ότι έχει θετική επιρροή. Κατάλαβα αυτά που είπατε. Χαιρετίζω τα σχόλιά σας και την προσέγγισή σας γενικότερα. Και σας ευχαριστώ και σας uh, Κύριε Σεβάγιο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Όντως αναφέρατε κάποια σημαντικά θέματα για την ανάπτυξη. Να σας διαβεβαιώσω ότι όποιο και αν είναι το αποτέλεσμα ε, για την ε, αναπτυξιακή βοήθεια, σίγουρα ελπίζουμε, όπως κατέστησε φέση και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι ό,τι και αν γίνει δεν θα είναι εις βάρος της αναπτυξιακής βοήθειας. Δεν θέλουμε να διώξουμε την ευθύνη από πάνω μας. Βέβαια, η ανάπτυξη ικανοτήτων είναι κάτι που θα συνεχίσει να μας απασχολεί και κύριε Πρόεδρε, ένα σχολείο σε αυτά που είπατε. Πιστεύω πως ε, φυσικά οποιαδήποτε ανταπόκριση θα πρέπει να είναι συνολική και να μην περιορίζεται μόνο στην Αφρική. Αλλά πέρα από αυτή και στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, στο Αφγανιστάν και σε άλλα μέρη. Και ο λόγος για τον οποίο είναι τόσο σημαντικό αυτό είναι ότι αυτό το μέσο συνδέεται με το Ευρωπαϊκό Ταμείο για την Ανάπτυξη. Βέβαια, ε, τούτων λεχθέντων, αν καταφέρουμε να μεγιστοποιήσουμε την ε, χρήση του μέσω αυτού στην Αφρική, στο μέλλον ίσως θα μπορέσουμε να εξετάσουμε και τη δυνατότητα χρησιμοποίησης άλλων μέσων. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριοι για την παρουσίασή σας. Για το ότι ήρθατε εδώ, πέμπτη, Πρωτού, θα, κλείσω τη συνεδρίαση θα ήθελα να συζητήσουμε τα διάφορα. Λοιπόν, δεν βλέπω κάτι στα διάφορα. Επόμενη συνεδρίαση, 16 Ιουνίου, 3 το απόγευμα, μέχρι τις 6.30 το απόγευμα και 17 Ιουνίου, πάλι από τις 3 μέχρι τις 6.30 το μεσημέρι. Σας ευχαριστώ πολύ και γεια σας.